αν εγκριθούν θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, αλλά φαίνεται πως έτσι θα τις αποφύγουμε. Θα υπάρχει συνεχώς κάποιος ο οποίος θα πληρώνει και θα υπάρχει ηθικός κίνδυνος. Εμείς λοιπόν είμαστε κατά. Ο κύριος Κλούτε έχει τον λόγο.